από τη ε, μαγνητοφώνηση ή τη ε, μαγνητοσκόπηση. Δεν ξέρω αν αυτοί οι αστεισμοί και ε, οι προκλήσεις έχουν θέσει στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την υπόδειξη αυτή. Θα δώσουμε την αντίστοιχη συνέχεια και θα δούμε τι συνέβη. Ευχαριστώ πολύ. So, machen wir weiter in der Tagesordnung. Συνεχίζουμε στη μέση διάταξη. Επόμενο θέμα είναι... Leichtfried για την αεροπορική ασφάλεια. Ο κύριος Λάιχτ Φρίντ ως εισηγητής έχει το για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η ασφάλεια στους εθέρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πάρα πολύ επίκαιρο θέμα. Εμείς δεν έχουμε καταφέρει να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και πληρώνουμε ένα τίμημα σε σχέση με αυτά. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο η πρόταση εκθεσής μου έχει σαν στόχο να αλλάξει η κατάσταση. Τι ακριβώς πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να σας πω εξ αρχής ότι θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους γιατί υπάρχει μια γενική θέληση από όλους να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια. Τι σημαίνει διαφάνεια. Από τη μια μεριά στο μέλλον οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να είναι σε θέση να δίνουν να παίρνουν καταρχήν τις πληροφορίες ώστε να είναι σαφές για τις αεροπορικές εταιρείες τι προβλέπεται σε βάση των προδιαγραφών ασφάλειας για αυτές και το επόμενο βήμα το οποίο αναφέρεται για τους, στους ίδιους τους επιβάτες είναι ότι μπορούν, θα μπορούν οι εταιρείε να πραγματοποιούν αυτά τα οποία προβλέπονται από τους κανονισμούς πτήσεων και ασφαλείας ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τηρείται απόλυτα η διαφάνεια σε αυτά τα θέματα ένα σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να τονίσω είναι το εξή ότι υπάρχουν πολλαπλά και διαφορετικά συστήματα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πτήσεων. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου πληρώνει το κράτος, αλλού πληρώνει ο καταναλωτής και μόνο, ο επιβάτης. Σε άλλα υπάρχει μεικτό σύστημα. Και γενικά πιστεύουμε ότι πρέπει τα συστήματα αυτά να παραμείνουν ως έχουν. Εμεί δεν πρόκειται να υπαγορεύσουμε σε ένα κράτο μέλο με ποιο τρόπο θα χρηματοδοτήσει τα συστήματα ασφάλειας των πτήσεων. Αυτό είναι δικό του θέμα. Υπήρξαν και διαφορετικές απόψεις σε σχέση με το ποιοι αερολιμένες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο, στην εμβέλεια αυτού του νομοθετήματος. Αλλά εδώ μιλάμε για ασφάλεια, δεν μιλάμε για κέρδη, δεν μιλάμε για τζίρο ή οτιδήποτε τέτοιο. Και επομένω η άποψή μα είναι ότι όλοι οι αερολιμένε οι οποίοι έχουν εμπορικέ πτήσει θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Αυτή νομίζω ότι είναι η σωστή άποψη. Και απόφαση. Τρίτον, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου υπάρχει μια μεγάλη ομοφωνία στην Ολομέλεια ότι θα πρέπει να κάνουμε μια σαφή διάκριση μεταξύ των τελών που έχουν να κάνουν για την εφαρμογή μέλων ασφαλείας που είναι πια τμήμα του κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λεγόμενων πιο αυστηρών μέτρων, τα οποία είναι μέτρα τα οποία προέρχονται εκ των έξω. Μπορεί ένα κράτο μέρο να κάνει ό,τι θέλει πέραν του κανονιστικού πλαισίου, αλλά αν εκφεύγει από το κανονιστικό πλαίσιο, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί το μέτρο αυτό από το ίδιο το κράτο μέλο. Χωρί καμία ε, χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκρίνουμε οποιοδήποτε μέτρο ασφαλεία χωρί να ξέρουμε ότι είναι πράγματι απαραίτητο. Θα πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό για του επιβάτε, τι σημαίνει για του αερολιμένε, τι σημαίνει για τι αεροπορικέ εταιρείε. Και εξάλλου θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα πριτανεύσει μια αρχή στην περίπτωση αυτή ότι η ασφάλεια είναι ένα καθήκον των δημοσίων φορέων. Δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο τις αεροπορικές εταιρείες, αφορά τα κράτη από τα οποία προέρχονται αυτές οι αεροπορικές εταιρείες και επομένως καταρχήν θα πρέπει να είναι στα χέρια των δημοσίων αρχών η ασφάλεια των αεροπορικών πτήσεων, επομένως και η χρηματοδότησή της. Είχαμε πάρα πολλές τροπολογίες, τρεις στον αριθμό. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλά τεκμηριωμένες. Υπάρχουν δύο πράσινες τροπολογίες τις οποίες εγώ θεωρώ ότι είναι άξιες να υποστηριχθούν. Η κυρία Λίχτεμπεργκε που είναι δίπλα μου μπορεί να μην συμφωνεί, αλλά νομίζω ότι τονίζουν την ανάγκη να τηρηθούν οι κοινωνικές προδιαγραφές οριελμένες, επομένως είναι απαραίτητο αυτό να το λάβουμε υπόψη όταν υπάρχει πραγματική πίεση κατά των αερολιμένων αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η κοινωνική διάσταση των εργαζομένων. Γι' αυτό θέλω να σε ευχαριστήσω αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ο κύριος Πίμπαλξ έχει το λόγο Κυρία Πρόεδρε, αγαπητά και έντιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Η πρόταση οδηγίας για την ασφάλεια των αεροπορικών πτήσεων είναι ένα τμήμα τη προοπτική μα για περισσότερη καινοτομία και ασφάλεια στον τομέα αυτό. Έχουμε ανερχόμενο κόστο ε, ασφάλεια λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων τη 11 η Σεπτεμβρίου 2001 και λόγω τη δημιουργία ενό κανονιστικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια των πτήσεων. Η νομοθετική αυτή πρόταση τη Κομισιόν έχει σαν στόχο να δημιουργήσει διαφάνεια και έλλειψη διακρίσεων στο κανονιστικό αυτό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τα τέλη ασφάλειας πτήσεων. Γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν θεωρεί ότι η ασφάλεια των πτήσεων και τα τέλη που απορρέουν από αυτήν θα πρέπει να καθορίζονται σε διαβούλευση με τους χρήστες των αεροδρομίων και πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα σε σχέση με το κόστος και την αποτελεσματικότητά του. Ο κύριο Λάιχτφριντ έκανε μια εξαιρετική εργασία ω εισηγητή. Θέλω ευχαριστήσω και όλα τα μέλη τη Επιτροπή Μεταφορών τα οποία συνέβαλαν σε αυτό το νομοθέτημα. Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση κινείται ακριβώ προ την κατεύθυνση <clears throat> την οποία θέλησε να ακολουθήσει και η Κομισιόν και υπογραμμίζω και δέχομαι και υπογραμμίζω μάλλον την υποστήριξη που δίνει στην Κομισιόν. Θέλω να σταθώ σε δύο μονάχα συγκεκριμένα θέματα τα οποία αναφέρονται και στην έκθεση του κυρίου Λάιχτφριντ. Καταρχήν η έκθεση του κυρίου Λάιχτφριντ εισαγάγει ένα νέο στοιχείο σε σχέση με ένα θέμα το οποίο είναι πολλές φορές αφιλεγόμενο. Ποιος θα πληρώσει την ύφη της αεροπορικής ασφάλειας. Η Κομισιόν λοιπόν έχει αντιμετωπίσει την άρνηση των κρατών μελών να αναλάβουν υποχρεώσεις και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο στη χρηματοδότηση της ασφάλειας στις πτήσει. Επομένως θα πρέπει να ακολουθήσουμε την αρχή της επικορικότητας και να αφήσουμε στα κράτη-μέλη καταρχήν να ρυθμίσουν τα θέματα αυτά. Επομένως με όλα αυτά μπορώ να, ε, <clears throat> να πω ότι η Κομισιόν υποστηρίζει αυτή την τροπολογία αλλά η τροπολογία 32 που αφορά τα κράτη-μέλη τα οποία χρηματοδοτούν περαιτέρω αυστηρότερα μέτρα, αυτό είναι κάτι το οποίο θα οδηγήσει ίσως σε έντονες συζητήσεις στο Συμβούλιο. Νομίζω όμως το γνωρίζει αυτό ο εισηγητής και περιμένει ότι θα υπάρξει και μια αψημαχία με το Συμβούλιο για τα θέματα αυτά. Επίσης, το θέμα της πιστοποίησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να εφαρμοστεί σε μέτρα τα οποία εκφεύγουν του κανονισμού αυτού. Αλλά πρέπει να σας πω ότι έχουμε ήδη κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι λειτουργούν και δεν θα πρέπει να τους ανατρέψουμε. Καταρχήν υπάρχουν οι ομάδες ε, συμβουλευτικού χαρακτήρα των εμπλεκομένων που αφορούν τους εκπροσώπους των, όλου του αεροπορικού κλάδου και που έχουν απόλυτα εμπλακή στη συζήτηση όλων των μέτρων για την αεροπορική ασφάλεια. Επίσης έχουμε και μια διαδικασία εποπτείας η οποία εξασφαλίζει ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του άρνηση κυρίας εάν το θεωρήσει ότι είναι απαραίτητο. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την τόσο εξαίρετη αυτή έκθεση και προσβλέπω στο να υπάρξει η έγκρισή του και να υπάρχει η έγκρισή της και να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Χάνς Πίτερ Μάρτιν. Συγγνώμη πρέπει να σας ενοχλήσω και πάλι, αλλά είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω σε ένα προσωπικό σχόλιο. Είναι χαρακτηριστικό. Άμα ζει κανείς στην Αυστρία, τα ξέρει αυτά. Υπάρχει μια ομάδα η οποία θέλει να μας βάλει μια ταμπέλα ότι είμαστε δεξιοί, ριζοσπαστικοί ακροδεξιοί. Τα άτομα αυτά δεν θέλουν να γίνεται η επιλογή των βουλευτών από τους, ε, από τους ε, πολίτες και αρνούνται οποιαδήποτε επαφή με μας. Αλλά διακόπτεται ο... Αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τι ακριβώς είναι η... ο χαιρετισμός του Χίτλερ μπορούν να καταλάβουν ποια είναι η πραγματικότητα. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά ως ε, δεξιό κόμμα και πρέπει να κάνω απόλυτα σαφές ότι εμείς είμαστε δημοκράτες. Αυτοί που είναι πραγματικά ακροδεξιοί κάθονται λίγο πιο έξω. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια σημαντική συμμετοχή στα τεκτενόμενα του Κοινοβουλίου. Δεν είμαστε ακροδεξιοί. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο αγωνίζεται για μεγαλύτερη δημοκρατία και δεν θέλει να είναι ακροδεξιό, δεν θέλει να είναι κοινικό και μισανθρωπικό κόμμα το οποίο αξίζει να πηγαίνει στους ψυχιάτρους και όχι στα κοινοβούλια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συζητήσουμε τη συζήτηση. Είναι διαδικαστικό? Παρακαλώ, διαδικαστικό. Υπάρχει και το θέμα στα 30 δευτερόλεπτα σηκώνουμε το γαλάζιο χαρτάκι. Θέλω να υποβάλουμε ερώτημα και αφορά τον προηγούμενο μιλητή. Δεν επιτρέπεται να κάνετε τέτοιε παρατηρήσει ε, με βάση την μπλε κάρτα. Γι' αυτό ε, ακυρώνεται η, η, η παρέμβασή σα. Ένα διαδικαστικό για ποιο άρθρο του κανονισμού. Εκτό μικροφώνου δεν ακούμε η παρέμβαση αυτή είναι απόλυτα αποδεκτή, η οποία όμως ε, διακόπτει μια συζήτηση για ένα συγκεκριμένο θέμα. Θα πρότεινα αυτά τα θέματα να συζητιώνται ανάμεσα στις συζητήσεις για τις εκθέσεις. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Την ε, προσωπική δήλωση την επέτρεψα επειδή Ε, επειδή το διαδικαστικό θέμα που ε, αναφέρθηκε πριν ε, αναφερόταν στον Hans Peter Μάρτιν, θα συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτηση τώρα για το θέμα μας και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει το λόγο ο κύριος Σαζάτα για δύο λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον εισηγητή, διότι η δουλειά του είναι πραγματικά έξοχη και η συνεργασία υπήρξε άριστη όταν επεξεργαστήκαμε από κοινό αυτό το έγγραφο. Έπρεπε να απαντηθούν τέσσερα ερωτήματα, αλλά πρώτα απ' όλα να καθοριστεί ένα καθήκον. Βασικό καθήκον ήταν να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των χρηστών των αεροπορικών εταιριών. Και αυτό ήταν ο βασικό μα στόχο. Και τέσσερα άλλα ζητήματα που θέσαμε ε, ήταν τα εξή. Διαφάνεια πάνω απ' όλα. Ποιε είναι οι ομάδες που μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Μετά, το εύρο, το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Ποια αεροδρόμια μπορούν να συμπεριληφθούν. Τρίτο το σημείο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε στο ερώτημά μας. Ευχαριστώ τον εισηγητή, διότι βρήκαμε μία λύση όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Ε, πρόκειται, πρόκειται περί αυστηροτέρας προσεγγίσεως. Πρέπει τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν στη χρηματοδότηση. Και μετά η διαχείριση και ο ανεξάρτητος φορέας όσον αφορά τον καθορισμό των τελών και των εισφορών όσον αφορά την ε, ασφάλεια των αερομεταφορών. Καταλήξαμε σε κοινή θέση. Είναι μεγάλη πρόκληση και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το Συμβούλιο. Ε, πιστεύουμε ότι η θέση μας, παρά το γεγονός ότι εγώ προσωπικά σαν επιβάτες πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να συνεισφέρουμε στις εισφορές, στα τέλη που καταβάλλω για την ασφάλεια, εν συγκρίση μάλιστα με άλλα μέσα μεταφορών. Λέω λοιπόν ότι οι επιβάτες των αεροπορικών εταιριών δεν θα πρέπει να ε, καταβάλουν κάποιο τίμημα για την ασφάλεια. Τούτου λεχθέντος όμως δεχτήκαμε μια συμβαστική θέση και θεωρούμε ότι ένα τέτοιο συμβιβασμό θα πρέπει επίση να υπάρχει από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Αλκαντράη για δυόμιση λεπτά. Συνάδελφοι, επίτροπε, αγαπητά μέλη, ευχαριστώ τον εισηγητή. Είναι έξοχο το έργο που επετέλεσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και όλους όσους συμμετείχαν στην προσπάθεια. Θα θυμόσαστε ότι το πρόβλημα της χρηματοδοτήσεως δεν είναι κάτι καινούριο Παιδευόμαστε με αυτό το ζήτημα από καιρό, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2001. Μιλήσαμε για μέτρα ασφαλείας και τότε. Ευθύς εξ αρχής το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε τη χρηματοδότηση και είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και θα πρέπει να εξευρεθούν πανευρωπαϊκές λύσεις. Δυστυχώς το Συμβούλιο ε, κόλλησε, αντιστάθηκε και δεν προχωρήσαμε. Να σας το υπενθυμίσω αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω το Συμβούλιο να ε, τηρήσει τις συμφωνίες του παρελθόντος. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια ειδική συμφωνία. Θα ήθελα να ζητήσω να τηρήσουν τη συμφωνία και να συνεργαστούν και να βρούμε μια εφαρμόσιμη λύση. Υπάρχουν διάφορες στοιχές που είναι σημαντικές. Η πιο ουσιαστική είναι η διαφάνεια. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ποιος πληρώνει το λογαριασμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που θέλουμε είναι να καταλήξουμε σε κάποιες συμφωνίες, να δοθούν υποσχέσεις και όταν δίδονται υποσχέσεις να τηρούνται. Αυτό πρέπει να γίνει. Οποιαδήποτε τέλη για την ασφάλεια που πληρώνονται θα πρέπει να πηγαίνουν στο συγκεκριμένο σκοπό και να μην χρησιμοποιούνται οι πόροι για κάτι άλλο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεύτερον, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα Θέλουμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ μέτρων ασφαλείας, επί των οποίων μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι μαζί, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και άλλων μέτρων, συμπληρωματικών μέτρων ασφαλείας που θέλουν να λάβουν τα κράτη-μέλη. Η διαφάνεια είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι εναπόκειται στα κράτη-μέλη να επομιστούν το οικονομικό βάρος θα πρέπει να πληρώσουν οι αδίποτε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Αλλά είναι περισσότερο κίνητρο αυτό για να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ευρωπαϊκό συντονισμό των μέτρων ασφαλείας. Και αν ληφθεί μια απόφαση όσον αφορά του σώματος σώματο κλπ., τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πληρώσουν το κόστο. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ για ε, την ομάδα Άλτε. Η κυρία Μάισνα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να, σας, να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Λάιχφριντ ε, και εκ μέρου ε, τη ε, κυρία Πράσια που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Συμμετείχε και αυτή στι διαπραγματεύσει και ήταν απόλυτα ικανοποιημένη η ποιότητα της ε, έκθεσης ε, φαίνεται και από το ότι στην ε, Επιτροπή η ψηφοφορία έβαλε ομόφωνο αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο το θέμα των καταναλωτών εδώ πέρα, είναι και η ασφάλεια στις ενέργειες μεταφορές. Θέλουμε να υπάρχει ασφάλεια και θέλουμε οι καταναλωτές να γνωρίζουν τι πληρώνουν και γιατί. Τα συστήματα αυτά είναι, διαφέρουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλος και δεν θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό, δεν θέλουμε να βιαστούμε. Θέλουμε όμως να υπάρχει διαφάνεια σχετικά με την ε, ανάλυση των δαπανών και ε, να γνωρίζει ο καταναλωτής τι πληρώνει. Αυτό δεν συμβαίνει πάντα μέχρι τώρα. Αυτό σημαίνει θέλουμε να ξέρουμε πόσο μεγάλο μέρος ε, του εισιτηρίου που υποτίθεται ότι είναι για την ασφάλεια πράγματι πηγαίνει για την ασφάλεια στις εναέριες μεταφορές δεν θέλουμε να βγάζει κανείς χρήματα από το θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ λογική ε, η θέση που έχουμε ε, διαμορφώσει. Υπάρχει ε, ένα βασικό θέμα όπου υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και στα κράτη-μέλη. Ποιο πληρώνει για την πρόσθετη ασφάλεια που, που αποφασίζεται, αυτό που θέλουμε στην Ευρώπη δηλαδή. Και αυτό τα κράτη-μέλη θεωρούν ε, ότι δεν πρέπει να πληρώσουν ε, παρότι το θέμα της εθνικής ασφάλειας είναι ε, εθνική υπόθεση. Το, το θέμα είναι θέλουμε σε σαρωτές σώματος, θέλουμε ε, κάτι τέτοιο να εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή όχι και ποιος θα πρέπει τελικά να πληρώσει και φυσικά θα πρέπει να πληρώσουμε. να, να αναρωτηθούμε κάτι τέτοιο θα επιφέρει περισσότερη ασφάλεια. Τέλει λοιπόν για την ασφάλεια στην η πρόεδρος ε, διακόπτη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φώστερ δεν είναι παρούσα. Έχει το λόγο η κυρία Ρόσπαχ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάποτε τα αεροδρόμια ήταν κάπου όπου αγόραζε κανεί ε, εισιτήριο, έδινε τι αποσκευέ του, ε, έδειχνε το διαβατήριό του και ε, πετούσε. Τώρα πια τα αεροδρόμια έχουν γίνει πόλει με ένα σωρό εγκαταστάσει, ταυτόχρονα όμω έχουν γίνει και Fort Knox με μέτρα ασφαλεία τα οποία πηγαίνουν προ μία κατεύθυνση. Έχουμε όλο και περισσότερα μέτρα. Και ναι, είχαμε ατυχήματα το παλιό καιρό, έχουμε και σήμερα και γι' αυτό είναι σημαντικό να ισχύουν μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τα ίδια μέτρα. Θα πρέπει να έχουμε ε, διαφανείς κανόνες για ε, τα αεροπλάνα και αυτό ισχύει για όλο τον κόσμο. Όλοι και οι επιβάτες και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τι καλύπτουν τα τέλη για την ασφάλεια. Κανένας δεν θα πρέπει να χάνεται σε μια ζούγκλα ε, τελών. Ο ε, καταναλωτή θα πρέπει να ξέρει ακριβώ σε τι καλύπτουν ε, τα τέλη αυτά. Δεν θα πρέπει να πηγαίνουν τα χρήματα αυτά. Στηρίζω απόλυτα την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Τελείωσε ο χρόνο σα, λέει η πρόεδρο. Προχωράμε στους επόμενους ομιλητές. Πρώτος έχει το λόγο ο κύριο Γκρό για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή για την εργασία που έχει κάνει. Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσε συζητήσει μαζί του από τι άλλε πολιτικέ ομάδε μαζί του στην Επιτροπή Μεταφορών, αλλά καταφέραμε να έχουμε ήδη συν... καταλήξει σε πολλέ συμβαστικέ λύσει σε ένα θέμα το οποίο στο παρελθόν ήταν πολύ αφιλεγόμενο και φαινόταν δεν υπήρχε περιθώριο για τέτοιε συμβαστικέ λύσει. Εμεί λοιπόν <clears throat> περιμένουμε την υποστήριξη τη Κομισιόν για να μπορέσει να υπάρξει μια ε, γενική αντιμετώπιση για τα τέλη το, της ασφάλειας για τις αεροπορικές ε, ε πτήσεις και όλα τα αεροδρόμια και όχι μόνο αυτά τα οποία πραγματικά ξεπερνάνε ένα όριο 5 εκατομμυρίων επιβατών. Είναι απαραίτητο να υπάρχει όμως από απόλυτη διαφάνεια για το ποιος πληρώνει, με ποιο στόχο και όλα αυτά και αυτό θα αφορά και, τις, ε, και τα αεροδρόμια, τη διαφάνεια και τις αεροπορικές εταιρείες. Γι' αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Αρχόμαι πάντα στο τρίτο σημείο που είναι το επίμαχο σημείο. Ποιο θα πρέπει να πληρώσει σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση. Εγώ πιστεύω ότι η δημόσια ασφάλεια πρέπει να καλυφθεί από δημόσια κονδύλια. Είναι ήδη μια ε, συμβιβαστική λύση με το να χρησιμοποιούμε την επικουρικότητα αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο όταν δεν βρίσκει κανείς λύση μαζί με το Συμβούλιο, καταλήγει στην επικουρικότητα. Αυτό δεν με ευχαριστεί ιδιαίτερα, αλλά τουλάχιστον αυτό το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι ότι οποιαδήποτε περαιτέρω μέτρα, πιο αυστηρά μέτρα, σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να καλύπτονται από τις δημόσιες αρχές. Τα τέλη ασφάλειας και η ασφάλεια γενικά έχει γίνει πολύ πιο πολυδάπανη το τελευταίο καιρό. Πρέπει να δούμε και την οικονομική πτυχή αυτού του θέματος σε ορισμένε περιπτώσει φτάνει το 12-13% του κόστου. και όταν μιλάμε λοιπόν για το τέλο, θα πρέπει να το σκεφτόμαστε αυτό ε, υπόψη μα. Τονίζω λοιπόν ότι θα πρέπει εμεί να διατυπώσουμε οι αιτήσει μα, μάλλον προ το Συμβούλιο και την Κομισιόν να έχουν κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Κύριε Τικάου για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η, η πρόταση αυτή προσπαθεί να θέσει ένα πλαίσιο για να καθοριστούν οι εισφορές για την ασφάλεια των αερομεταφορών. Και είναι ένα σύστημα που δεν οδηγεί στη διακρίση. Η ασφάλεια στα αεροδρόμια είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αλλά στο τέλος οι επιβάτες είναι εκείνοι που πληρώνουν μέσω των εισιτηρίων που αγοράζουν μέσω πληρώνουν για τα μέτρα ασφαλεία. Γι' αυτό θα πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτε ξεχωριστά ποιο είναι το κόστο ασφάλεια που συμπεριλαμβάνεται στην τελική τιμή. Ε, αυτή η οδηγία και η οδηγία που αφορά τα τέλη των αεροδρομίων, οι δύο οδηγίες θα πρέπει να εναρμονιστούν. Ζήτησε επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτές τις οδηγίες τα τέλη που αφορούν την ασφάλεια των αερομεταφορών να χρησιμοποιούνται από τους φορείς των αεροδρομίων για να θέτουν, να εφαρμόζουν μέτρα ασφαλείας αποκλειστικά. Επιπλέον το Κοινοβούλιο ζήτησε διαφάνεια αυξημένη όσον αφορά αυτά τα τέλη. Τα κράτη-μέλη δίνανται όμως να επιβάλλουν πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας αν το επιθυμούν, αλλά το κόστος θα πρέπει να καταβληθεί από τα λόγω κράτη-μέλη. Τα μέτρα ασφαλείας δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τη ροή των επιβατών στα αεροδρόμια. Δυστυχώς, κυρίως το αεροδρόμιο των Βρυξελών, αντιμετωπίζουμε ουρές, ατέρμονες ουρές επιβατών που περιμένουν για να μπορέσουν να περάσουν από τον έλεγχο ασφαλείας και να ταξιδέψουν. Ε, παρομοίως θα ήθελα να αναφερθώ στην απαγόρευση κάποιων υγρών που απαγορεύεται να μεταφερθούν εντός του αεροσκάφους και επιτρέπεται να κατασχεθούν κάποια προϊόντα. Και δυστυχώ, στο αεροδρόμιο των Βρυξελών, παραδείγματο χάρη, υπάρχει μια πολύ επαχθή διαδικασία που οδηγεί στην κατάσχεση κάποιων προϊόντων. Είναι μια διαδικασία που δυστυχώς δεν επιτρέπει να υπάρχει δυνατότητα στο τέλος, στον προορισμό, να ξαναβρει κανείς τα προϊόντα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τικάου. Έχω μια ερώτηση μπλε κάρτας. Ε, θέλετε να απαντήσετε. Παρακαλώ κύριε Όπερμαγερ. Θα ήθελα να διορθώσω. Ενώ σε τη διαδικασία catch the eye. Ωραία, ναι. Μερικέ φορέ η μπλε κάρτα έχει δύο σημασίε. Ωραία, καμία ερώτηση. Catch the eye. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Προχωράμε τώρα. Ο κύριο Πάσκα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τα τέλη ασφάλεια είναι πρόσθετο κόστο για τι αεροπορικέ εταιρείε και τα αεροδρόμια τα οποία μετακυλίονται άμεσα στους χρήστες, δηλαδή στους επιβάτες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξεύρουμε μηχανισμούς οι οποίοι θα αποφύγουν η προσθέμενη αξία μέσα σε εισαγωγικά που θα έπρεπε να είναι το τέλος ασφάλειας να μην είναι ένα πρόσχημα για ορισμένου οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν περισσότερα χρήματα με το πρόσχημα της πρόσθετης ασφάλειας. Το τέλος ασφαλείας θα πρέπει να έχει σαν στόχο πραγματικά αποκλειστικά και μόνο να εξασφαλίσει την ασφάλεια των επιβατών. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μονάχα με μέτρα τα οποία θα είναι διάφανα, με μέτρα και κανόνες που θα μπορέσουν στο μέλλον να διευκολύνουν την ε, σωστή λειτουργία των ε, μέτρων ασφαλείας και δεν θα επιτρέψουν σε αεροπορικές εταιρείες να αυξάνουν αλόγιστα το κόστος των αεροπορικών ναύλων και επίσης να αυξάνονται και τα διάφορα τέλτα που επιβάλλονται. Εμείς θα πρέπει να μην δημιουργήσουμε νέους φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς προσθέμενη αξία. Θα πρέπει να έχουμε μονάχα φορείς οι οποίοι βοηθούν τον Ευρωπαίο πολίτη. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ένα κάπως διευρυμένο λεπτό. Τώρα ξανά θέτουμε το χρονόμετρο στο 0 και ελπίζω ότι υπάρχει αρκετό χρόνο για όλου, Δύο λεπτά κύριε Σμέλτσα. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Λόγω τη έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία υπήρξαν δεκάδε χιλιάδε πτήσεων οι οποίε ακυρώθηκαν. Αυτό είναι ήδη μία ένδειξη του τι σημαίνει η ασφάλεια των πτήσεων. Ποιος θα πληρώσει όμως για μια τέτοια φυσική καταστροφή και σε ποιο βαθμό ήταν δικαιολογημένες οι απαγορεύσεις πτήσεων. Δεν είναι μονάχα θέμα των Υπουργών Μεταφοράς. Θα πρέπει και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσουμε ποιο είναι το κόστος το οποίο πρέπει να επιμείνεται ο επιβάτης σε σχέση με τις περιοριστικές, τα περιοριστικά αυτά λεγόμενα αντιτρομοκρατικά μέτρα. Γιατί δεν πιστεύω ότι μπορεί να μετακυλεί κανείς το κόστος ασφάλειας απλώς στον πολίτη και στον καταναλωτή θα πρέπει να αποφύγουμε να υπάρξουν χρήσεις μέτρων όπως οι σαρωτές πλήρου σώματος και η αφαίρετη χρήση τέτοιων εργαλείων. Εμείς μέσα σε συμφωνίες όπως η SWIFT δίνουμε τη δυνατότητα να δώσουμε δεδομένα στις ΗΠΑ για τους πολίτες μας και στις αρμόδιες αρχές τους. Αυτό όμως δεν η συζήτηση που κάνουμε δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη την επιβάρυνση, την αυξανόμενη επιβάρυνση των εναρίων ελεγκτών που έχουν τεράστιο φόρτο εργασία. Υποτίθεται ότι η, ότι η αλλαγή προς ένα ενίο σύστημα εφαίρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μείωνε το, το κόστος και θα είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Δεν έχει επιτύχει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Βλέπουμε λοιπόν πόσο εύκολα μπορεί να υπάρξει ένα χάος, εναέρειες μεταφορές, απλώς και μόνο από την έκρηξη ενός ηφαιστείου. Κύριε Ντεβεράκ, για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα συγχαρώ τον εισηγητή μα, τον κύριο Λάχτριτ, για το κείμενό του και για το πνεύμα συνεργασία που επέδειξε στο θέμα. Υποστηρίζω κυρίω αυτά που αφορούν τι προτάσει του όσον αφορά τη χρηματοδότηση τη ασφαλεία των αερομεταφορών, διότι εδώ μιλάμε για αυτό το θέμα και όχι, την, ε, και όχι κάτι άλλο. Εδώ και πολλά χρόνια η, Ευρωπαϊκή, Επιτροπή μα πολεμάει για να γίνει αποδεκτή αρχή σύμφωνα με την οποία τα αυστηρότερα μέτρα όσον αφορά τα θέματα ασφαλεία θα πρέπει να τα πληρώνουν τα κράτη-μέλη και υποστηρίζω πλήρω τον εισηγητή από αυτού. Η ασφάλεια δεν αφορά μόνο του επιβάτε αλλά όλου του πολίτε και είναι ευθύνη των κρατών μελών να λάβουν τα μέτρα εκείνα κατά πολεμήσεως τη τρομοκρατία Άρα δεν δικαιολογείται οι επιβάτες των αεροπορικών εταιριών να είναι μόνοι εκείνοι που πληρώνουν για το κόστος των μέτρων ασφαλείας στα αεροδρόμια και επί των αεροσκαφών. Και στους σιδηροδρόμους και στις θαλάσσιες μεταφορές βλέπουμε ότι τα κράτη κατά περίπτωση εν μέρη εξ ολοκλήρου χρηματοδοτούν τα μέτρα ασφαλείας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στεναροί εναντί του Συμβουλίου και να υπερασπιστούμε την τροπολογία 32 μέχρι τέλους της ε, εκθέσεως που υθετήθηκε την Επιτροπή Μεταφορών. Θα ήθελα να άλλο σε άλλο σημείο ακροθυγό. Αν υποστηρίζω τι προόδου που πετεύχθησαν όσον αφορά τη μη διάκριση και τη διαφάνεια που θα επιφέρει το κείμενο, ε, δεν πιστεύω ότι στόχο τη εν λόγω οδηγία είναι να τεθεί σε εφαρμογή ευρωπαϊκό σύστημα ενίο και ταυτόσιμο όσον αφορά τι εισφορέ για την ασφάλεια, τα τέλη για την ασφάλεια. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν κοινοί κανόνε, αλλά επιτρέπεται και στα κράτη-μέλη να κρατήσουν τα παρόντα συστήματα όσον αφορά την ίσπραξη των τελών και σε κράτη όπω είναι η Ισπανία, η Ιταλία ή η Γαλλία, όπου τα τέλη ψηφίζονται από το Κοινοβούλιο και αντί αυτή περιπτώσει θα πρέπει η αρχή, αρχή προσφυγής κατά του νόμου που θα πρέπει να είναι η αρχή εποπτείας. Και αυτή είναι, αυτός είναι ο στόχος της τροπολογίας 40 που ελπίζω να υποστηριχθεί από πολλούς όταν θα την ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί η κυρία Άγια Σέντερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε παρά τις δυσκολίες που ήταν απόλυτα ανάγλυφες αυτή τη βδομάδα σε σχέση με την έλλειψη ενιαίων εθέρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ότι δεν υπάρχει μια ενιαία αρχή για τον έλεγχο και την εποπτεία των εθέρων, σιγά σιγά αρχίζουμε και προχωρούμε στο στόχο αυτό και το κείμενο αυτό είναι ένα περαιτέρω πετραδάκι και εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή. Ο κύριος Λάιχτφριντ αξίζει κάθε επένου για το έργο του και για την ε, αντιμετώπιση την θετική που είχε για τα θέματα της ασφάλειας και, των, και τα κοινωνικά θέματα. Ίσως είμαστε υπερβολικά μαξιμαλιστικοί και ξεχνάμε ότι το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Είναι χρήσιμο να έχουμε ένα κοινό σύστημα με ανεξάρτητες αρχές, με διαφάνεια σε σχέση με τα τέλη και όλα αυτά, να σεβόμαστε το περιβάλλον και τα κοινωνικά θέματα, αλλά Νομίζω η Κομισιόν να μπορέσει να, μου διευκρινίσει καλύτερα αν υπάρχουν κάποια στοιχεία, κάποιες ψηφίδες που ελείπουν. Όπως είπε η κυρία Δεβεϊράκ, δεν υπάρχει αναγνώριση μέσα στο σύστημα ενός τρόπου με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει αυτά τα τέλη με συμφωνία κοινοβουλευτικού χαρακτήρα και υπάρχει ο φορέας αυτός ο οποίος τα εφαρμόζει. Τι βιωσιμότητα μπορεί να έχει τέτοιο κείμενο όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές μεταξύ ημών και του Συμβουλίου και του γεγονότος ότι δεν υπάρχει συμβατότητα κατά την άποψή μου μεταξύ αυτού του εγγράφου και της οδηγίας για τα τέλη στους αερολιμένες. Υπάρχει μια τεράστια λοιπόν αβεβαιότητα η οποία πλανάται σε σχέση με το ποιο θα πληρώσει το κόστος αυτής της ασφάλειας που δέχομαι ότι πρέπει να είναι δημόσιου χαρακτήρα αλλά όταν λέμε τα κράτη σε τελική ανάλυση δεν είναι τα κράτη κάτι το αφηρημένο, είναι οι φορολογούμενοι οι οποίοι πληρώνουν. Είμαστε εμεί οι οποίοι ταξιδεύουμε σε τελική ανάλυση. Πιστεύω λοιπόν ότι η Κομισιόν θα έπρεπε να μα πει ποια είναι η άποψή του για το πώ βλέπει το μέλλον αυτού του κειμένου και τι θα μπορέσει να ευδοκιμήσει από αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Μαρινέσκου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πράγματι οι αρωματοφορές είναι το πιο, ο πιο ασφαλής τρόπος μεταφορών και όλα αυτά τα γεγονότα σε αερομεταφορές μπορεί να έχουν ε, διεθνείς συνέπειες, όπως είναι η δεκαήμερη διακοπή των πτήσεων λόγω της εκρήξης του ηφαιστείου. Θα πρέπει να, ε, να δούμε ποιος είναι στα λυσίδα. Είναι οι αεροπορικές εταιρείες, ε, τα αεροσκάφη, οι επιβάτες, τα αεροδρόμια. Είναι μια λυσίδα στον τομέα τη ασφάλεια και θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ των τομέων επικοινωνία χωρί να υπάρχουν σφάλματα. Ανησυχεί ο επιβάτη για την άνεσή του, για το ταξίδι του και δεν καταλαβαίνει πάντα ότι τα μέτρα ασφαλεία είναι απόλυτα αναγκαία. Και ίσω να μην καταλαβαίνει ότι αυτό συνεπάγεται και κόστο. Ο επιβάτη δεν ξέρει κάποια δράματα που λαμβάνουν χώρα. Δεν γνωρίζει ακριβώ ποιε ήταν συνέπειε τη ε, επίθεση τη 11 Σεπτεμβρίου. Τι γίνεται με αν κάνει ένα σφάλμα ο πιλότο, αν υπάρχει παρεξήγηση επικοινωνία μεταξύ πιλότου και πύργου ελέγχου, αν υπάρχουν απρόβλεπτε ατμοσφαιρικέ συνθήκε. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη την ασφάλεια. Χρειάζονται σαφή μέτρα που να μπορούν να εφαρμόζονται, να εφαρμόζονται και να εφαρμόζονται κατά γράμμα οι κανόνε. Συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε εξαιρετικά μέτρα σε κάποιε περιπτώσει. Αυτό αναφέρεται στην έκθεση. Αλλά αυτά τα μέτρα θα πρέπει να είναι διαφανή. Οι επιβάτε έχουν το δικαίωμα και θα πρέπει να μπορούν να ε, αντιμετωπίζουν διαφάνεια, διαφανή μέτρα και να ξέρουν την αλήθεια. Δυστυχώ η διαφάνεια επικοινωνία στον τομέα τη αεροπορική, τη ασφαλεία σε αερομεταφορέ χρειάζεται βελτίωση. Και αυτό είναι καθήκον των αεροδρομίων, των αεροπορικών εταιριών που θα πρέπει να δείξουν μεγαλύτερη διαφάνεια. Οι επιβάτε, σε αντάλλαγμα, θα πρέπει και αυτοί να καταλάβουν ποια μέτρα ασφαλεία στα αεροδρόμια και στα αεροσκάφη, ακόμα και αν είναι δυσάρεστα και δεν είναι άνετα, ουσιαστικά είναι απαραίτητα και είναι προ όφελό του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σούλμερ, για δύο λεπτά. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Λάχτφριντ για την εξαιρετική του έκθεση η οποία ε, μεταφέρει ένα πολύ καλό περιεχόμενο. Ποιο είναι το θέμα μας τελικά. Είναι το θέμα η ασφάλεια, η προστασία του καταναλωτή, ε, ο συντονισμός, ε, η διασφάλιση της ποιότητας. Και αναφέρεται το θέμα της δημιουργίας μιας νέας αρχής που θα ασχολείται με τα θέματα αυτά. Βρίσκω θετική την επικουρικότητα στην έκθεση και θα πρέπει να διατηρηθεί για μένα σημαντικό είναι να υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στα τέλη και στους φόρους ε, και ε, θα Πρέπει ε, όλες οι σχετικές αρμοδιότητες, ε, οι αστυνομικές, ε, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας κτλ. θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από φόρους, όχι από τέλη των χρηστών. Είναι θέματα που ενδιαφέρουν τα κράτη-μέλη και έχουμε και τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να ληφθούν και στον τομέα αυτό στο θέμα αυτό θα πρέπει όποιος ε, αναθέτει τις αρμοδιότητες αυτές ε, στις αρχές ε, να πληρώνει και για αυτές. Θα πρέπει λοιπόν να δηλώνουμε μονοσήματα περί τίνος πρόκειται εδώ πέρα. Όσον αφορά την μελέτη αντικτύπου που μας έχει υποβάλει η Επιτροπή, αναφέρεται συμβολή 0,1% για τις δαπάνες αυτές. Δεν θα πρέπει να ξεκινήσουμε πολύ ψηλά. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ε, καταλήξουμε σε έναν καλό συμβασμό και με την ε, ε, Ομοσπονδιακή Γερμανία που έχει ιδιαίτερε ανησυχίε όσον αφορά την επικουρικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ερχόμαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος, κύριε Βολτορόφ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υποστηρίζω απόλυτα αυτή την πρόταση γιατί βελτιώνει σημαντικά τη διαφάνεια των τελών <clears throat> και των ε, ποσών τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί δεν υπάρχει μια προσπάθεια να επιτύχουμε ένα υψηλότερο επίπεδο εναρμόνισης. Ίσως λόγω της κυρίαρχης θέσης ορισμένων αεροδρομίων οι επιβάτες πληρώνουν υπερβολικά τέλη τα οποία δεν οδηγούν σε καλύτερη ταχύτητα ελέγχου ασφαλείας ή πιο αποτελεσματικά μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια αυτά. Πριν από δύο χρόνια εφαρμόστηκε η οδηγία και η Κομισιό θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη και να προτείνει να υπάρχει ένα ενιαίο τρόπο για τον υπολογισμό των τελών ασφαλεία. Συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε ε, σε ορισμένε περιπτώσει πιο πολυδάπανα και αυστηρά μέτρα όπως οι σαρωτές πλήρου σώματο, Αυτό όμω πρέπει να καλύπτονται οικονομικά από τα κρατημέρια και όχι από του επιβάτε. Εγώ αναρωτιέμαι για το πώ μπορούν να ερμηνευθούν αυτά τα τέλη ασφαλεία από τα αεροδρόμια ή από τις εταιρείε που αυξάνουν το κόστος στον άβλο. Κύριε Πάσκο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Λάιχτφριντ έχει δίκιο. Οι δαπάνες για την επιπλέον ασφάλεια θα πρέπει να καλύπτεται τελικά από τα κράτη-μέλη. Άλλωστε, οι επιβάτες ως πολίτες ούτως ή άλλως πληρώνουν τα κράτη-μέλη για την ασφάλειά τους. Δεν μπορεί το κράτος να λέει στους πολίτες του ότι θα πάρετε ε, ότι επιπληρώσατε. Η υποχρέωση των κρατών προχωράει πέρα από αυτό διότι το κράτος δεν είναι απλά άλλος ένας ε, παρόχος υπηρεσιών που με μοναδικό κίνητρο το κέρδος. Ε, σας θυμίζω την απλή αυτή αλήθεια διότι παρά την αρχή αυτή οι επιβάτες και όχι τα κράτη πληρώνουν τελικά το λογαριασμό για την αυξημένη ασφάλεια όπως πολύ σωστά σημειώνει ο εισηγητής. Επιπλέον, ε, πολύ συχνά η επιπλέον ασφάλεια που, ε, ε, από την οποία αποφελούνται οι επιβάτε που παρέχεται από, όχι από τα κράτη αλλά από επιχειρήσεις και αυτό δεν είναι σεβασμός των δικαιωμάτων των επιβάτη. Θα πρέπει να σταματήσει η πρακτική αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Όμπερμα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε καθότι το θέμα των τελών για την ασφάλεια στην ε, πολιτική αεροπορία ε, είναι αντικείμενο διαφορετικού χειρισμού στα, διάφορα, στα διαφορετικά κράτη-μέλη, ε, βρίσκω πολύ σημαντικό να υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στα τέλη αυτά και στις υπηρεσίες που παρέχονται και θα πρέπει να οριστούν σαφώς αυτές και θα πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής γιατί πράγμα πληρώνει. Θα πρέπει να γίνεται κατανοητό πώς ε, υπολογίζονται τα τέλη αυτά. Το ύψος δηλαδή και η φύση των τελών αυτών θα πρέπει ε, να εξηγούνται σαφώς, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Θα πρέπει να αποφύγουμε ε, τη στρέβλωση του ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αυτοί ήταν ε, οι ομιλητέ στη διαδικασία Catch the Eye. Τον λόγο έχει πάλι η Κομισιόν. Παρακαλώ, κύριε Επίτροπε Πίμπαλξ. Πρόεδρε, μέλη, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και όσον αφορά την ασφάλεια των αερομεταφορών, όλοι έχουμε τις εμπειρίες μας. Θα μπορούσα να αναφέρω και δική μου εμπειρία ε, ε, και δεν με αφήσαν να μεταφέρω κάποια πράγματα όπω τη ΡΗ. Ε, νομίζω ότι όμως παρόλα αυτά έχουμε βελτιώσει το σύστημα ασφαλεία. Η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπής προχωράει ένα βήμα πιο πέρα, διότι αν υπάρχει ασφάλεια υπάρχουν τέλη και ο πρώτο κανόνα είναι διαφάνεια. Πιστεύω ότι η έκθεση και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενισχύουν το ένα το άλλο. Όσον αφορά το ποιο τελικά αναλαμβάνει το κόστο, η άποψή μου είναι ότι η επικουρικότητα είναι η καλύτερη λύση, διότι ούτω ή άλλω δεν είναι τα κράτη-μέλη, οι πολίτε είναι εκείνοι που πληρώνουν. Το μόνο ερώτημα είναι, θα είναι ότι όλοι οι φορολογούμενοι ε, θα πληρώνουν ή οι επιβάτε. Αυτό δεν είναι απλό ερώτημα να απαντηθεί και γι' αυτό νομίζω ότι στην πρότασή μα η επικουρικότητα έλαβαν υπόψη τις ισχύουσε διευθετήσει. Το Κοινοβούλιο προχωρά πιο πέρα και βλέπει όλο τον τομέα τη ασφάλεια των αερομεταφορών. Θα δούμε που θα μα οδηγήσει η συζήτηση, αλλά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια αξιοπρεπέστατη πρόταση και χαίρομαι πάρα πολύ που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν γέννη δέχεται την πρόταση και ανεβάζει τον πύχη ω συνήθω της προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να δούμε που θα οδηγηθούμε αλλά πιστεύω ότι η πρότασή μας υπευλήθη εγκαίρως και καλύπτει το σωστό πεδίο εφαρμογή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πίμπαλξ, κύριε Επίτροπε και πάλι ο εισηγητής, ε, σύντομο κύριε Λάιχτ και Φρίντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να παρατείνω ιδιαίτερα τη συζήτηση. Θέλω να χρησιμοποιήσω όμως αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω και εγώ τους σκιώδεις εισηγητές από όλα τα κόμματα οι οποίοι και αυτοί εργάστηκαν πάρα πολύ κυρία Λίχτεμπεργκ, ο κ. Κόλτσικ, ο κ. Ζασάδα και άλλοι. Εδώ και ένα χρόνο ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα, κάναμε πολύ μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική στα θέματα αυτά ομού. Και ένα δεύτερο θέμα, θέλω να ευχαριστήσω το Συμβούλιο, αλλά να κάνω και μια έκκληση προς το Συμβούλιο. Η Επιτροπή Μεταφορών είναι μια επιτροπή που θέλει να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά με ψυχραιμία και αντικειμενικότητα. Παρ' όλα αυτά ήρθαμε σε σύγκρουση με το Συμβούλιο. Εμείς έχουμε δείξει τη θέλησή μας να προχωρήσουμε σε συμβασμούς. Δεν πρέπει όμως το Συμβούλιο να ξυπνά κύονες οι οποίοι υπνώτουν. Δεν πρέπει λοιπόν το Συμβούλιο να έχει μια στάση η οποία είναι άκαμπτη και δεν έχει καμία πρόθεση να δεχτεί τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τότε αυτό θα προκαλέσει μια αντίδραση από τη δική μου Επιτροπή. Και το είπαν και ορισμένοι συνάδελφοι. Αν το Συμβούλιο δεν θέλει να προσεγγίσει τις απόψεις του Κοινοβουλίου, εμείς δεν θα δεχτούμε ούτε τους σαρωτές πλήρου σώματος, ούτε πολλά άλλα από τα μέτρα τα οποία θέλει να προωθήσει το Συμβούλιο. Αυτό δεν είναι προς το γενικό συμφέρον δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να συμβεί και γι' αυτό σας παρακαλώ να σκεφτείτε λίγο καλύτερα τα κράτη-μέλη δεν μπορεί να θεωρούν ότι μετά από την έγκριση συνθήκης της Λισαβόνας δεν μπορεί να, αντιμετωπί... μπορεί να αντιμετωπίζουν στο Κοινοβούλιο. Θυμηθείτε το SWIFT. Ευχαριστώ. Έχει κλείσει η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει στην επόμενη Σύνοδο Ολομέλειας στις Βρυξέλλες. Και τώρα Ερχόμαστε στο επόμενο σημείο.